την κυρία Γιουστίνα Βιτκαουσκάιτε από την 21η Νοεμβρίου 2012 και την κυρία Μόνικα Παναγιώτοβα από την 6η Δεκεμβρίου 2012. Προτείνω αυτές ε, οι εντολές ε, να ακυρωθούν. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Η κύρωση ε, εδόθη και ισχύουν οι εντολές αυτές. Από την αρμόδια ομάδα έχω αιτήματα από